Φεβρουαρίου 2015. Απευθύνω χαιρετισμό πρώτα στον Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κύριο Ντόναλτ Τούσκ και του δίνω ευθύ αμέσω το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε. Σας ευχαριστώ. Ξέρω κύριε Βουλευτέ, Πρόεδρε Γιούγκερ, με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ ξανά στο Κοινοβούλιο, ένα μήνα μόλι μετά τη συνάντηση του Συμβουλίου. Ε, γιατί το Συμβούλιο Κορυφής έχει ως ε, στόχο όχι τις διαπραγματεύσεις αλλά τη διαβούλευση. Και γι' αυτό και επομένω είναι συγκεκριμένα τα αποτελέσματα. Οπότε το πλαίσιο που κινηθήκαμε ήταν οι ταχείες εξελίξεις. Ε, είδαμε ποιε δεν οι προκλήσεις προς συζήτηση. Η πρώτη πρόκληση ήταν η Ουκρανία. Με τον Ποροσέγκο, τον πρώτο της χώρας, είχαμε ανταλλαγή απόψεων, ο οποίος ήρθε στο Συμβούλιο για να μας παρουσιάσει τη συμφωνία του Μίντ και να μας πει πώς βλέπει τα πράγματα ε, εκεί. Η Αγία Μέρκελ επίσης ε, κατέβαλε κάποιες προσπάθειες απαραίτητες για την επίτευξη της ε, ειρήνης. Το ίδιο ισχύει και για τις πρωτοβουλίες της Νορμανδίας και τις σχετικές συνομιλίες. Τελικά έκλεισε κάποια συμφωνία, πάρα πολύ όμως, αλλά η Ένωση ακόμη ελπίζει ότι θα υπάρξει κάποια ειρήνη που θα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και εδαφική κυριότητα της χώρας. Και αυτό θα γίνει σύντομα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε ακόμη πολύ επιφυλακτικοί. Η συμφωνία του Μίνσκ του 2014 δεν τηρήθηκε. Οι ηγέτες συζήτησαν για το πώς θα εφαρμόσουν τη συμφωνία, αλλά εάν δεν την εφαρμόσουν, τότε και εμείς χωρίς δεγμό θα αναλάβουμε δράση. Η δέκατη του πυρός υποτίθεται ξεκίναγε 15 Δευτέρου τα μεσάνυχτα. Όμως παραβιάστηκε πάνω από 800 φορές σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΕ. Είμαι σε συνέχεια επαφή με τον πρόεδρο Λόντ, ε, κυρία Μέρκελ και όλους τους ηγέτες, γιατί είμαστε ενωμένοι στο θέμα της Ουκρανίας ακόμη βρίσκονται και εκκρεμούν προς επιπλέον κυρώσεις. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τις ευχάριστες ή δυσάρεστες εξελίξεις. 12 Φεβρουαρίου είχαμε την τρομοκρατική απέσια απόπειρα που είχε αυτά τα θύματα και οπότε είπαμε ότι τώρα θα καταρτήσουμε ένα αντιτρομοκρατικό πρόγραμμα. Και αυτό ε, το περιλάβαμε στην κοινή δήλωση κατόπιν της συνάντησης κορυφής Οπότε τώρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι ήδη κάνει και να το συνεχίσει όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια. Όμως θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα και να τα κάνουμε ταχύτερα. Δηλαδή, να εκμεταλλευτούμε τους μηχανισμούς του Σαγγεν καλύτερα, ίσως να αναθεωρήσουμε τους ε, κανονισμούς για τους ε, συναγερμούς ε, πυρκαγιάς κλπ. Είδατε επομένω ότι με αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις δείξαμε το πώς είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε κάθε εξτρεμισμό και κάθε είδος τρομοκρατία. Και με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι είμαστε απολύτως αλληλέγγυοι προς την Δανία, τον λαό της Δανίας, αλλά και τις οικογένειες των θυμάτων στο άτιμο Συμβούλιο Κορυφή δεν συζητήσαμε μετά τη Λιβύη. Όμω είχαμε εκεί πέρα αποτρόπαια τρομερά γεγονότα σε αυτή την ε, χώρα. Οπότε βεβαίω και πρέπει να ασχοληθούμε. Γιατί η εθνική ασφάλεια είναι θέμα εθνική κυβέρνηση. Όμω υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί τομεί όπου μπορεί ο ένα να στηρίξει τον άλλο και οπότε και επιβάλλεται ανάληψη κοινή δράση. Οπότε και σε σχέση με αυτό θεωρώ πολύ θετική την πρόοδο που είχαμε για επανεκκίνηση των ε, συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το PNR τα στοιχεία των επιβατών, οπότε έτσι θα έχουμε περισσότερη προστασία των πολιτών, αλλά χωρίς να θίξουμε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Οπότε και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι όλοι να βάλουμε ένα χεράκι, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει σχετικό τον Ιούνιο και για άλλα πράγματα. Πάντως, στο μεταξύ, νυφάλια, όλοι μαζί, θα αντιμετωπίσουμε τις απειλές και με αποφασιστικότητα. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα. Η συνάντηση του Φεβρουαρίου δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή, ούτως ώστε να έχουμε κάποιο είδους ασυντόνιστες διαπραγματεύσεις για το πρόβλημα της Ελλάδας. Αλλά είχαμε τον ε, πρόεδρο του Eurogroup που ήρθε να μας πει πώς έχει κατάσταση των πραγμάτων όσον αφορά τις επαφές με την ε, Ελλάδα. Επίσης ήρθε και ο Πρωθυπουργό ε, Τσίπρας, νέο μέλος του Συμβουλίου, ο οποίος και αυτός μας εξέθεσε το πώς βλέπει τα πράγματα. Και συμφωνήσαμε ότι οι συνομιλίε θα συνεχιστούν. Έτσι και έγινε. Θα συνεχιστούν σε υπουργικό επίπεδο τόσο ώστε να βρεθεί ένα κοινό παρονομαστής. Αναμφίβολα, έτσι πίστευα ότι θα γίνει από πριν. Οπότε χρειάζεται στενή επαφή με όλα τα μέρη, όλου του εμπλεκομένου, τόσο ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια σύμφωνια και είδατε τι έγινε στο Eurogroup τη Παρασκευής. Οπότε, και εγώ περιμένω πώ και πώ να δω πώ οι υπουργοί θα δώσουν το πράσινο φω όσον αφορά τα ε, προγράμματα μεταρρυθμίζουν τη Ελλάδα. Αυτό το οποίο είναι χθε. Οπότε, είδαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για Οικονομική και Ένωση. Θα πρέπει βέβαια η χάραξη πολιτικής να βελτιωθεί και θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη διαμόρφωση. Πάρα πολύ σημαντικό ότι ξεκίνησε μια τέτοια προβληματική. Ο δε πρόεδρος Γιούγκερ μα παρουσίασε μια ανάλυση και ε, απήντησε σε κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν να θέλουμε να πετύχουμε καλύτερη οικονομική διαχείριση. Τώρα κάτι άλλο το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί. Μετά την προσφατή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι προτεραιότητες ήταν ούτως ώστε να μπορέσουν οι εθνικές οικονομίες να είναι πιο συμβατές με την νομισματική ένωση. Αυτό όμως πώς θα γίνει. Θα γίνει μόνο με ισχυρό βολονταρισμό σε εθνικό επίπεδο. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα κοιτάμε μπροστά, στο επόμενο Συμβουλίο. Τι επόμενε τρει εβδομάδε πρόκειται να παρακολουθήσουμε τι εξελίξει και σε Ουκρανία και σε Λιβύη. Μέρα προ μέρα, με μεγάλο ενδιαφέρον. Και τον Μάρτιο η συνάντηση κορυφή πρόκειται να είναι η ώρα χάραξης πολιτικής προς Ανατολάς και προς Νότον. Να δούμε τι θα γίνει και με την ευρωπαϊκή οικονομία, γιατί βέβαια θα πρέπει να εστιάσουμε προσοχή μας σε κάτι το οποίο προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά ενδιαφέρει πάρα πολύ και πολλούς βουλευτές. Ότι δηλαδή πήγη εξέβρεση λύσεις για την Ενεργειακή Ένωση, ακριβώς όπως ο κύριος Σεύκοβιτς προλίγου σας ανέλησε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να σημειώσει πρόοδο και σε αυτό το μέτωπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Θα ακολουθήσει ο Πρόεδρος Γιούνκερ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Συμβούλιο της 12 η Φεβρουαρίου ήταν ένα άτυπο Συμβούλιο. Δεν ελήφθησαν αποφάσεις δηλαδή. Ήταν ένα χρήσιμο Συμβούλιο και παρά τα όσα είχαν ακουστεί νωρίτερα, ήταν ένα συμβούλιο χωρίς δράματα. Σύντομο, αποτελεσματικό, όπως και ο πρόεδρος του. Φυσικά, μερικές εβδομάδες μετά τα γεγονότα του Παρισιού συζητήσαμε για την τρομοκρατία και από αυτού θέλω να πω ότι συμφωνήσαμε η συμφωνία, ότι η συμφωνία Σέγγεν δεν δημιουργεί πρόβλημα. Η Συμφωνία Σέγγεν είναι η απάντηση στο πρόβλημα. Γι' αυτό και αποκλείσαμε, βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε ιδέα να προχωρήσουμε σε σημαντικές και ουσιαστικές τροποποίησεις της Συμφωνίας Σέγγεν. Όταν πρόκειται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δεν πρέπει να δρούμε βιαστικά, βεβιασμένα. Η απάντηση στην τρομοκρατία δεν μπορεί να γίνει στα βιαστικά. Α θυμηθούμε τα σφάλματα των Αμερικανών φίλων μας, τι κάνανε αμέσως μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον. Πρέπει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, όντας βέβαια σοβαρή. Και αυτό ακριβώς κάναμε όσον αφορά το PNR. Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω το Σώμα που συμφώνησε με την ε, απόφαση μιας κοινοβουλευτικής σας επιτροπής. Και σας θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, διότι το Κοινοβούλιο, οι κοινοβουλευτικές του επιτροπές, τα οργανά του, οι ευρωβουλευτές μπόρεσαν και προσέγγισαν στη θέση της προηγούμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από τη δικιά μου. Δεν επικρίνω το Κοινοβούλιο για την απόφαση που είχε πάρει πριν από μερικούς μήνες, διότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων φυσικά είναι ε, πράγματα ε, τα οποία σέβεται πολύ και, το και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα πρέπει να δρούμε πάντα με ηρεμία. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του Συμβουλίου συζητήσαμε και για την ενέργεια. Σήμερα το πρωί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε μια απόφαση για αυτό το θέμα. Εγώ πάντα θεωρούσα ότι στην αρχή της θητείας πρέπει να αρχίζουν τα μεγάλα σχέδια. Δεν το έκανα αυτό πάντα στη ζωή μου. Ίσως αν το είχα κάνει και νωρίτερα, τα αποτελέσματα να ήταν προτιμότερα και καλύτερα. Τώρα όμως θέλω να ξεκινήσουμε με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη από την αρχή. Γι' αυτό και συμφωνήσαμε πράγματι επί μιας πράσινης βίβλου όσον αφορά την ε, ενιαία αγορά κεφαλαίων. Ξέρω ότι δεν συμφωνούν όλοι. Μπλε βίβλο. Καλά, αυτό εξαρτάται που τοποθετείται κανείς. Ο Φιλίπ προτιμάει την πράσινη βίβλο βέβαια. Αλλά το θέμα είναι οι απαντήσεις που θα δώσουμε να είναι και αυτές πράσινες. Τέλος πάντων, η αυτοψία θα δείξει, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την Ενεργειακή Ένωση, όπως σας είπα. Και φροντίσαμε για τη διαφάνεια, τη μεθοδολογία ε, της Επιτροπής και τα λοιπά, να ξεκαθαριστεί αυτό, πώς δηλαδή θα προχωρήσουμε και πώς θα δουλέψουμε. Σκοπεύω να υιοθετήσω κάθε απόφαση που χρειάζεται λοιπόν για να προχωρήσουμε και στην ψηφιακή αγορά. Το Μάιο θα γίνει αυτό. Όλα τα μεγάλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν μπήκανε στο αυλάκι και πολύ σύντομα θα ξέρουμε περισσότερα. Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου λοιπόν, υπό την Προεδρία του Πρόεδρου Τίσκο, παρουσιάσαμε μια αναλυτική μελέτη για τις αιτίες της κρίσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Και μια που ήταν το πιο εύκολο, απαριθμίσαμε στους συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές ερωτήσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της ΟΝΕ. Μου είπαν ότι θα έπρεπε να διαβάσω εδώ ότι ορισμένοι ε, δεν χάρηκαν που μόνο ερωτήσεις είχα. Ναι, αλλά αν δεν έχω ερωτήσεις δεν μπορώ να έχω και απαντήσεις. Εγώ θέλω οι απαντήσεις να ανταποκρίνονται στις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση. Θα αντεξετάσουμε λοιπόν όλα αυτά και με τον πρόεδρο Τισκ και με τον πρόεδρο Ντάισελπλουμ και με τον πρόεδρο Τράκη μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα συνεργαστούμε όσο γίνεται πιο στενά και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτού. Θέλω επίσης να διευκρινίσω ότι πρόκειται για έκθεση τεσσάρων προέδρων. Και ο Μάρτιν Σούλτς δηλαδή θα συμμετέχει. Δεν είναι μία έκθεση των τεσσάρων θεσμικών οργάνων συν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι προσωπική δουλειά του καθενός από εμά. Οπότε όπως έκαναν και οι υπόλοιποι πρόεδροι μέχρι τώρα θα πω και εγώ ότι θα εξετάσουμε τις προσωπικές μας ιδέες, όχι των θεσμικών μας οργάνων. Εγώ είχα βέβαια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν έγινε συζήτηση στο Συμβούλιο. Ο κύριος Ντράγκη επίσης είναι σε ένα ανεξάρτητο όργανο. Δεν ξέρω τι έκανε. Εμείς πάντως πρέπει να ξέρουμε ότι πρόκειται για τις προσωπικές απόψεις των πέντε πρόεδρων. Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχει και αυτός σε αυτό το εγχείρημα. Όσον αφορά τώρα το επενδυτικό πακέτο, δεν ξέρω αν είναι σωστό το όνομα ή όχι, πάντως με να μ' αρέσει. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις κοινοβουλευτικές του επιτροπές και τους δύο εισηγητές που δουλεύουν πάνω σε αυτό για το εξαιρετικό τους έργο, τον κύριο Μπούλμαν και τον κύριο Φερνάντες, οι οποίοι με το έργο τους θα επιτρέψουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει για το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα και για το νομοθετικό κείμενο που θα το συνοδεύσει. Η απόφαση θα ληφθεί το αργότερο τον Ιούνιο. Πρέπει όντω να ληφθεί κοινοβουλευτική απόφαση μέχρι τον Ιούνιο. Και πρόεδρε, θέλω να πεθυμίσω εδώ ότι επιλέξαμε την κοινοτική μέθοδο για να εγκριθεί το κείμενο αυτό. Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφασίσει να αποφασίσει μόνη τη Επιτροπή ή το Συμβούλιο. Εγώ θέλησα και σας το είπα να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο, γι' αυτό και προτίμησα την κοινοτική μέθοδο. Και αυτήν ακριβώς πρέπει να εφαρμόσουμε για αυτό το θέμα. Επίσης, σήμερα, συλλογικά, το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε και για τις δημοσιονομικές πτυχές που έχουν να κάνουν με κάποιες χώρες μέλη. Όχι μία, πολλές χώρες μέλη. Και επειδή το κοινό αλλά και οι βουλευτές προσέχουν πάρα πολύ το τι γίνεται στη Γαλλία, Πρέπει να σας πω ότι σήμερα αποφασίσαμε ότι καλέσαμε την ε, Γαλλία να αναθεωρήσει το έλλειμμά της τώρα για το 2015 κατά 10,5% που σημαίνει ότι πρέπει να τροποποιήσει τον προπολογισμό που έχει ψηφίσει για το 2015 και να μειώσει το διαρθρωτικό του έλλειμμα γύρω στο 0,8-0,9%. Δώσαμε δύο χρόνια παραπάνω στην Γαλλία και αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που έχει να κάνει με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δηλαδή η Γαλλία θα είναι, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, υπό ενισχυμένη εποπτεία. Σημαίνει ότι πιο στενά θα συνοδεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Γαλλία όσον αφορά τις ε, διορθώσεις που θα κάνει τις δημοσιονομικές. Δουλεύουμε λοιπόν, εργαζόμαστε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα όσα επιθυμείτε να κάνουμε, αλλά για αυτά που κάνουμε βασιζόμαστε και στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Επιτροπή δεν μπορεί ούτε να μιλήσει ούτε να δράσει. Βασιζόμαστε σε εσά λοιπόν. Ο Πρόεδρος Σούλτς, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, προχωρούμε τώρα στη συζήτηση. Πριν όμως ανοίξουμε τη συζήτηση, δύο σύντομες ανακοινώσεις. Πρώτο, θα προσέχω επακριβώς την τήρηση του χρόνου. Γιατί μου το ζήτησαν και οι πολιτικές ομάδες να τηρηθεί αυστηρά το όριο του χρόνου αγορεύσεως. Γνωρίζετε ότι γενικά είμαι γενναιόδωρος, όμως στην περίπτωση αυτή είμαι υποχρεωμένος να τηρώ αυστηρότατα τα χρονικά όρια. Εξάλλου, δεν θα επιτρέψω ούτε τη χρήση των κιανών καρτών, ούτε και διαδικασία catch the eye. Δεύτερη ανακοίνωση, σημαντική αυτή, στα θεσμικά μας όργανα έχουμε τακτικά εξασκουμένους σταζιέρ. Οι ασκούμενοι αυτοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έπαιξαν ποδόσφαιρο κατά των ασκουμένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και σας λέω τώρα το αποτέλεσμα. 10 προς 1, 10-1 κέρδισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτό οφείλω να το πω εν παρουσία του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος σηκώνεται αμέσως. Είμαι σύμφωνος με το αποτέλεσμα, λέει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Κύριε Τούσκ, γνωρίζετε ότι είστε κι εσείς παλαιός ποδοσφαιριστής όπως και εγώ. Να φτιάξουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα και στο Συμβούλιο και να δούμε πόσοι ασκουμενοί σας θα τα καταφέρουν απέναντι στους δικούς μας. Τώρα, ακολουθεί εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο κύριος Σάριου Βόλσκι. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ. Κύριοι Πρόεδροι, Μόνο δύο εβδομάδες πέρασαν από το τελευταίο άτυπο συμβούλιο και μου φαίνεται σαν να πέρασαν αιώνες. Τόσο πολύ έχει επιταχυνθεί ο χρόνος. Το συμβούλιο αρχικά υποτίθεται ασχολούνταν με τρομοκρατία. Η ζωή έφερε άλλα δύο θέματα. Την Ελλάδα, την κρίση της Ελλάδας και την Ουκρανία υπό επίθεση. Αυτές οι τρεις υποθέσεις τι κοινό στοιχείο έχουν είναι δοκιμασία για τις ευρωπαϊκές αξίες. Πρώτο, για το ε, περιοδικό Σαρλί, τρομοκρατία, ασφάλεια των πολιτών. Εκεί σχέδιο δράσης, όπως εξήγησε ο πρόεδρος Τούσκ. Δεύτερο, Ελλάδα. Υποστηρίξαμε την τήρηση των συμφωνηθέντων. Ίδιοι κανόνες για όλους και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ταυτόχρονα όμως συνδυάσαμε την υπευθυνότητα αυτή με αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Και πρόεδρε Γιούνκερ, δεν τα κάναμε όλα όσα είχαμε υποσχεθεί απέναντι στην Ελλάδα. Τέλος, το τρίτο, Ουκρανία. Επίσης μεγάλη δοκιμασία και έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τις δύο προηγούμενες υποθέσεις. Το περιοδικό Σαρλί δηλαδή και την κρίση στην Ελλάδα. Πρόκειται για τρομοκρατία και πρόκειται και για οικονομική κατάρρευση στην περίπτωση της Ουκρανίας. Αλλάζουν τα σύνορα της Ουκρανίας με άσκηση βίας, με κρατική τρομοκρατία από τη Ρωσία και με διεξαγωγή πολέμου. Θα τηρήσουμε την πορεία, όπως είπε ο πρόεδρος Τούσκ, μιας εξωτερικής πολιτικής βασισμένης σε αξίες. Θα τηρήσουμε τις αρχές μας που λένε παραπάνω κυρώσεις εφού παραπάνω πόλεμος. Θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στο Κίεβο. να αντιμετωπίσουμε τον επιτιθέμενο αλλά να και υποστηρίξουμε και το θύμα σε, βασισμένη σε δύο αρχές του διεθνούς δικαίου. Πρώτο, δικαίωμα άμυνας. Δεύτερο, ευθύνη για την υποστήριξη. Για όλα αυτά όμως, για να γίνουν όλα αυτά, χρειαζόμαστε να είμαστε ισχυροί μέσα στην Ένωση. Ακολουθεί ο κύριος Πιτέλα, εξ ονόματος του ε, κόμματος των, της ομάδας μάλλον των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε Γιούγκερ, για αυτό που εξαγγείλεται δηλαδή αυτό το μέλλον για το μέλλον της Ευρώπης έγινε να προσυπογραφεί και από τους πέντε Προέδρους. Θα ήταν κατανοητό να μην προσυπογράψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούσε κανείς να το εξηγήσει κανέναν και θα ήταν και άδικο. Οπότε και θα πρέπει βέβαια να διδαχτούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μέσω του πρόεδρου μας πρέπει να βρούμε σε εξουσίες κατάστασης και πρώτα πρέπει να τοποθετηθούμε πρώτα πρώτα όσον αφορά την Ελλάδα. Η υπηρεχθήσα συμφωνία είναι κάτι το θετικό, οπότε θα πρέπει να εξηγηθεί σε όλους ότι σεβόμεθα το αποτέλεσμα των εκλογών. Είναι αδιανόητο να σκεφτόμαστε ρεβάνς σε σχέση με κάποια κυβέρνηση που έχει αναλάβει τα καθηκοντά τη. Μα αρέσει, δεν μα αρέσει. Αυτή είναι η κυβέρνηση επίση. Θα πρέπει να κατανοήσουμε το νόημα, το μήνυμα αυτών των εκλογών. Είναι μια αντίδραση αντίθετα με την λιτότητα. Οπότε τώρα θα πρέπει να λειτουργήσει αυτή η κυβέρνηση και θα πρέπει να περάσει από την φάση της προπαγάνδας ή στην φάση των επιλεγών όσον αφορά συγκεκριμένα διλήμματα. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή μεταρρύθμιση στα κοινωνικά, στα οικονομικά, η δημοκρατία τη διαφθορά, σε όλα αυτά. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να τύχουν απάντηση επίσης τώρα για την εξωτερική πολιτική. Ο πρόεδρο τους που μα παρουσίασε την κατάσταση, τον ευχαριστώ, ευάλωτη εκείνη η συμφωνία, αλλά καλύτερα από το τίποτα. Οπότε θα πρέπει να ενδυναμώσουμε την πολιτική μας, να πρέπει να πιέσουμε την Ρωσία, να κάνουμε ό,τι πέρα χέρι μας να κάνουμε, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια εκεχηρία η οποία να πιάσει τόπο και ε, ενδεχομένως να μετασχηματιστεί σε ειρήνευση, Λιβύη. Ευχαριστούμε Πρόεδρε τους και εσείς μας. Υπενθυμίσατε ότι υπάρχει και η Λιβύη η οποία αποτελεί ένα θέμα τραγικό, δραματικό, το οποίο δεν την χάνει επαρκούς προσοχή. Προέρχονται από εκεί τρομερή κίνδυνη για όλους. Επομένως και θα πρέπει και εμείς οπωσδήποτε να εστιάσουμε προσοχή μας εκεί. Όλα αυτά τα οποία μας είπε και η ε, κυρία Μογκερίνη. Τώρα όσον αφορά την μετανάστευση. Λαμπεντούζα. Είχαμε τον τρίτον τώρα, όπως θέλετε πέστε, τρίτον, τράιτον, αλλά ο τρίτονας που βρήκαμε δεν αρκεί. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε το Μάρε Νόστρομ που να είναι πραγματικά ευρωπαϊκός φορέας, οπότε καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας. Φυσικά κανένα πρόβλημα με το PNR, θα πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά δεν αρκεί το PNR, δεν αρκούν οι κατάλογοι με τα στοιχεία των επιβατών για δεδομένε τρομοκρατία. Θα πρέπει να κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα. Και επίση ε, εύχομαι να τα πετύχουμε. Ευχαριστούμε κύριε Πιτέλα. Και τώρα. Τι έχετε, ένα διαδικαστικό εσείς. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς όπως είπαμε και προηγουμένως. Μονομερός δεν δικαιούστε να τροποποιήσετε την εγκριθήσα ημερησία διάταξη. Την εγκριθέ στην αρχή της συνάντησης. Και είπαμε ότι μετά τη συζήτηση πρέπει να γίνει συζήτηση του τύπου Κάτς Διάε, πρόεδρος. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Μορβάη. Δεν δικαιούμαι να τροποποιήσω την ε, ημερησία διάταξη μονομερός Δεν το έκανα αυτό όμως. Έχουμε τη διάταξη 162, παραγράφη 6 και 7, που διέπουν τη διαδικασία με τις γαλαζιές κάρτες και το κάτι Και εκεί ορίζεται ότι οποτεδήποτε κατά τη συζήτηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γαλαζιές κάρτες. Όμως στην αρχή σας είπα ότι δεν έχουμε χρόνο για τέτοια πράγματα. Άρα το κάτσε και Οι κάρτες μπορούν να μόνο εάν υπάρχει χρόνο Οπότε για καθίστε και διαβάστε πάλι το 162. Και τώρα η κυρία Φωτίγκα από το ECR. Honorable President. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ονειρεύτηκα, ονειρεύτηκα την Ευρωπαϊκή Ένωση των ονείρων μου ακριβώς αλλά και των ελπίδων μου. Πίστευα ότι θα είχαμε να κάνουμε μία ανταλλαγή απόψεων και με τον εκπρόσωπο της χώρας η οποία έχει πέσει θύμα επίθεσης. Νομίζω ότι έχουμε τις αρμοδιότητες έτσι ώστε να αποφασίσουμε να διαπραγματευτούμε φοβαρά. Τώρα τι σημαίνει το λεγόμενο σχήμα της Νορμανδίας στην ουσία αυτό είναι έλλειψη παρουσίας εκπροσώπων του Συμβουλίου, της Προεδρίας του Συμβουλίου και ε, απουσία φυσικά της υπευθύνου για την εξωτερική πολιτική. Μια πάρα πολύ επιφυλακτική στάση γενικά ε, ακόμα και στα πλαίσια της ομάδας των 7 η στήριξη που δόθηκε ε, δεν ήταν η σωστή. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχουμε μία απλή σύγκρουση, έχουμε να κάνουμε με πόλεμο, έχουμε να κάνουμε με προσάρτηση, έχουμε να κάνουμε με παραβίαση εθνικής κυριαρχίας, έχουμε να κάνουμε με κατοχή και έχουμε να κάνουμε και με έλλειψη αποφασιστικότητας από πλευράς μας πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι η Ρωσία, η Ρωσική Ομοσπονδία σε καμία περίπτωση δεν τήρησε τα συμπεφωνημένα σχετικά με την Ουκρανία. Και όμως κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου αποφασίσαμε ότι δεν θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό. Σημαίνει ότι στην ουσία εμείς αφήνουμε να παγιωθεί η σύγκρουση αυτή. Empowering the EU Λοιπόν, ε, είναι σαφές ότι θα πρέπει να αλλάξουμε στάση και θα ήθελα η απόφαση του άτυπου συμβουλίου να μην είναι γενικού τύπου απλά πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα και στα πλαίσια της οδηγίας για το PNR. Στην πολιτική μου ομάδα έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό αναλυτικά. Τώρα, για την Ελλάδα υπάρχουν δύο πλευρές. Φυσικά ε, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στις συζητήσεις που έχουμε με τους λαούς της Ευρώπης για τις πιθανές συνέπειες της νομισματικής ένωσης. Θα πρέπει επίσης να μην ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι η αποδοχή της Ελλάδας ήταν μια πολιτική απόφαση. Όπως πολιτική ήταν η απόφαση και για την νομισματική ένωση και την ίδρυσή της και δεν μπορούμε να εμείνουμε αποκλειστικά στα οικονομικά χαρακτηριστικά. Ο Πρόεδρος Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για το PNR στον πρόεδρο Γιούγκερ. Κοιτάξτε, δεν, δεν είπαμε ότι θα παραιτηθούμε από τα δικαιώματά μας. Είπαμε ότι εμείς ψηφίσαμε κάτι το ξεκάθαρο. Θέλουμε ένα ευρωπαϊκό PNR, γι' αυτό ζητάμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάγκη της αναλογικότητας, που είναι βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός συστήματος και ζητάμε και από το Συμβούλιο να περάσει στην έγκριση της οδηγίας για τα, για τα προσωπικά δεδομένα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν είμαστε εμείς οι οποίοι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις θέσεις μας, θα πρέπει από κοινού τα τρία όργανα, εφόσον το Συμβούλιο κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και η Επιτροπή κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, τότε θα μπορέσουμε και εμείς να προχωρήσουμε. Μαζί θα το κάνουμε αυτό κύριε Πρόεδρε, όχι ο καθένας στο δικό του δρόμο. Τώρα για την οικονομική διακυβέρνηση. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε ένα καλό βαθμό. Ε, με αυτές τις συμβατικές ρυθμίσεις νομίζω ότι μας απασχόλησαν για πολύ καιρό και ότι δηλαδή η Επιτροπή θα έκανε μια ειδική συμφωνία με το κράτος μέλος για τις μεταρρυθμίσεις. Όχι, τα αφήνουμε αυτά τώρα. Πρέπει να περάσουμε σε μια σύγκληση γενική, ευρωπαϊκή, για την Ευρωζώνη και για την Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι ακολουθείτε τώρα τον σωστό δρόμο. Το τρίτο θέμα το οποίο συζητήθηκε για την Ελλάδα ήταν σοφή η απόφαση η οποία ελήφθη να δοθεί δηλαδή χρόνος τεσσάρων μηνών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συμφωνίας. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες μπορούν να περιγράψουν ε, ε, με σωστό τρόπο τις μεταρρυθμίσεις που θέλουν να κάνουν. Ήταν μια σοφή απόφαση. Ελπίζω να γίνουν ε, πραγματικές ρυθμίσεις στον τομέα της φοροδιαφυγής, στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Αυτά δεν επαρκούν ακόμα εγώ δεν έχω εντυπωσιαστεί αν θέλετε από την επιστολή της ελληνικής πλευράς εδώ και λίγες μέρες. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, το άνοιγμα των ε, επαγγελμάτων, ε, μείωση και μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα και αυτό είναι μια τεράστια ανάγκη. Και τέλος, θα πρέπει οι δημόσιες τράπεζες ή οι τράπεζες σε δημόσιο έλεγχο να γίνουν ε, τράπεζες ανταγωνιστικές στον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε τις επιπλέον λεπτομερέστερες προτάσεις από πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης πριν να ε, προχωρήσουμε. Ήταν λοιπόν μια σωστή απόφαση αυτή την οποία πήρατε να δώσουμε τέσσερις μήνες ε, στην ε, κυβέρνηση. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει συγκεκριμένε προτάσεις σε λίγες μέρες. Τώρα και έρχομαι τελικά στο θέμα της Ουκρανίας. Το είπατε 800 φορές ότι παραβιάστηκε η συμφωνία. Το είπατε και το ξαναλέτε, η συμφωνία Μίνσκ 2. Θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό. Αυτό σημαίνει η στρατηγική την οποία ακολουθούμε απέναντι στη Ρωσία είναι η σωστή στρατηγική. Ε, στην ουσία μπαίνει στην Κρυμαία η Ρωσία και εμεί αντιδρούμε εκ των υστέρων. Μετά μπαίνει η Ρωσία στις ανατολικές ε, επαρχίες της Ουκρανίας και εκ των υστέρων πάλι αντιδρούμε. Παραβιάζει ε, τη Συμφωνία Μίνσκ 2 και ίσως εδώ να αντιδράσουμε. Κοιτάξτε, όχι, δεν πρέπει να περιμένουμε. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε, τώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε για τις συμπληρωματικές κυρώσει, όχι αμέσως να τις εφαρμόσουμε, αλλά να πούμε ότι αν πράγματι συνεχίζεται να παραβιάζεται, τότε εμείς θα επιβάλλουμε τις εξή οικονομικές κυρώσεις. Όχι μόνο να καθόμαστε στην άκρη και να περιμένουμε και να αντιδρούμε εκ των υστέρων σε αυτά τα οποία κάνει ο Πουτίν. Θα πρέπει να αποφασίσουμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επί τη βάση των προτάσεων Μογκερίνη και Τάσκ ποιες θα είναι οι νέες οικονομικές κυρώσεις και να πούμε στην ηγεσία της Ρωσίας ότι αυτές οι κυρώσεις θα γίνουν πραγματικότητα αν συνεχίσετε σε αυτό το δρόμο τον επιθετικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει για την Ηνωμένη Αριστερά ο κ. Παδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απάντηση που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Eurogroup, η Κομισιόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα θέματα που έθεσε η ελληνική κυβέρνηση είναι και ένας καθρέφτης για το πώς θα αντιμετωπίσει τα ίδια τα δικά της τα προβλήματα η Ευρωζώνη. Γιατί αυτά τα χρόνια έχουμε μείωση των επενδύσεων στην Ευρωζώνη, οικονομική στασιμότητα, αποπληθωρισμό τον κίνδυνο μιας νέας ύφεσης, αύξηση της φτώχειας και της ανεργίας σε όλη την Ευρωζώνη. Υπάρχει μια μελέτη της McKinsey που λέει ότι στα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αύξηση του δημόσιου χρέους σε όλη την Ευρωζώνη. 15 από τα 19 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης έχουν χρέος πολύ πάνω από το όριο που έθεσε η συνθήκη του Μάστριχτ. Επτά από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης έχουν δημόσιο χρέος πάνω από 100%. Και τη μεγαλύτερη αύξηση του χρέους τα τελευταία χρόνια την έχουν οι τέσσερις χώρες που μπήκαν σε μνημόνια. Η Ιρλανδία 172% αύξηση του δημόσιου χρέους, η Ελλάδα 103% αύξηση του δημόσιου χρέους, η Πορτογαλία 100% αύξηση του δημόσιου χρέους και η Ισπανία 72% αύξηση του δημόσιου χρέους σημειώνω με ικανοποίηση ότι σήμερα η συζήτηση για την Ελλάδα δεν είναι στους πολεμικούς εκδικητικούς τόνους που υιοθέτησαν οι Γερμανοί χριστιανοδημοκράτες πριν λίγες ημέρες που θέλαν να εκδικηθούν τον ελληνικό λαό γιατί ψήφισε αντίθετα με τις δικές τους επιθυμίες. Σημειώνω θετικά τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Κομισιόν ο κύριος Γιούνκερ πριν λίγες ημέρες μιλώντας στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όπου είπατε κύριε Πρόεδρε, ότι φερθήκατε απαράδεκτα ως ευρωπαϊκή θεσμή απέναντι στους Έλληνες, τους προσβάλατε και ότι έγιναν και λάθη στην εφαρμογή του προγράμματος. Αυτό που δόθηκε με την απόφαση του Eurogroup δεν είναι μόνο μια χρονική ανάσα. Είναι η δυνατότητα να συνδυαστούν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η ανάγκη να τηρούνται οι κανόνες και το δεύτερο είναι η ανάγκη να σεβόμαστε όλη τη δημοκρατία και το αποτέλεσμα των εκλογών που λέει ότι κάτι πρέπει να δούμε, μήπως πρέπει να τα αλλάξουμε και κάναμε λάθος. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε, αποδεχόμενοι τις δεσμεύσεις μας και ζητάμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής ζητώντας και τεχνική βοήθεια κάτι που όπως είπε ακόμη και ο δόκτωρ Σόιμπλε αρνήθηκαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ζητάμε και την ενίσχυση του επενδυτικού πακέτου Juncker με κριτήρια όπου να κατευθυνθούν αυτές οι επενδύσεις στις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη γιατί έχουν μεγαλύτερη ενεργεία και μεγαλύτερη αποεπένδυση. Και φυσικά να αξιοποιήσουμε και την ευελιξία στο σύμφωνο σταθερότητας που ένας πρώην επίτροπος αρμόδιος για το θέμα ο κ. Πρόντι είχε χαρακτηρίσει ηλίθιο και την ποσοτική χαλάρωση που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κλείνω με δύο λέξεις για το θέμα της Ουκρανίας. Η ειρηνευτική συμφωνία είναι ένα μικρό δεντράκι. Κινδυνεύει να ξεραθεί. Η δουλειά η δική μας είναι να ενισχύσουμε με ψυχραιμία αυτή την ειρηνευτική προσπάθεια. Και για το θέμα της αντιμετώπισης των τρομοκρατικών επιθέσεων εκτός από την αλληλεγγύη μας στους λαούς της γαλλίας και της δανίας σημειώνω θετικά την ψύχρεμη τοποθέτηση του κυρίου Γιούνκερ ότι δεν πρέπει να κάνουμε τα λάθη που έκαναν οι Αμερικανοί μετά το 2001. Σας ευχαριστούμε και τώρα από τους πράσινους ε, το λόγο έχει ο κ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα βασικά να μιλήσω για την Ελλάδα και θέλω να αναρωτηθούμε. Χρειαζόμαστε όλο αυτό το ψυχόδραμα που έχει κρατήσει σχεδόν τέσσερις εβδομάδες. Με αυτό το ψυχόδραμα η ελληνική κυβέρνηση προσποιεί ότι ε, μετά τις 25 Ιανουαρίου διαρκούσε ακόμη η προεκλογική εκστρατεία και λέγαν «Α, στόχευσε η χώρα μας και ε, αυτό είχε επιπτώσεις από πλευράς ΕΚΤ. Επέμενε επίσης για το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Εξίσου ανεύθυνη ήταν ε, η αιμονή κάποιων μελών ε, του Συμβουλίου να λένε ότι θα το πληρώσει η Ελλάδα, θα βγει από την Ευρωζώνη η Ελλάδα, όπως τη δεκαετία του 20 με τη Γερμανία. Και είναι ανεύθυνο διότι ο Υπουργό Οικονομικών τη Γερμανίας, ο Wolfgang Σόιμπλε, ήταν ο πρώτος που το έκανε αυτό ε, και νομίζω ότι η χώρα του έχει τρεις φορές πτωχεύσει, τον προηγούμενο αιώνα δεν θα έπρεπε να μιλάει. Λοιπόν, έχουμε του τέσσερι μήνες τώρα, καλό είναι αυτό θα πρέπει να του χρησιμοποιήσουμε για να βρεθεί μια συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και του εταίρου τη. Τρία είναι τα βασικά σημεία αυτής της ε, νέας ε, συμφωνία. Ε, θα πρέπει να είναι βιώσιμο, να γίνει βιώσιμο το χρέο τη Ελλάδα. Στην ιστορία τη σύγχρονη οικονομία, ποτέ μια χώρα 4,5% του ΑΕΠ δεν το χρησιμοποίησε για την αποπληρωμή του χρέου. Εντάξει, Νορβηγία για δύο χρόνια. Και εδώ μιλάμε για μια 20 ετία στην περίπτωση της Ελλάδας. Λοιπόν, η εξυπηρέτηση του ε, χρέους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3,5% μακροπρόθεσμα και με άλλες βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις. Δεύτερο βασικό στοιχείο και επιμένω ότι είναι πολύ πιο αξιόπιστη η νέα κυβέρνηση σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, σε ΙΠΑΣΟΚ, ε, σε σχέση με την ε, ε, ε, θέσπιση ε, μιας φορολογικής μηχανής, φοροεισπρακτικής μηχανής στην Ελλάδα. Υπάρχει τεχνογνωσία και υπάρχει δύναμη κρούση σε σχέση με την Ελβετία, παραδείγματο χάρη, ώστε να έχουμε πληροφορίες και την υποβολή, καταβολή κάποιων οφειλόμενων φόρων. Τρίτο στοιχείο θα πρέπει η οικονομία να μπει ε, στον ε, δρόμο μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή είναι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, επενδύσεις, ενεργειακή μετάβαση, τα λέγαμε σήμερα. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει καθαρός εξαγωγίας ενέργειας προς τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδού λοιπόν μια πηγή, κατ' εμέ, ε, σημαντικού εισοδήματος για το κράτος και για την ελληνική οικονομία. Θα πρέπει λοιπόν να δειχθεί σε προτεραιότητα ε, η επένδυση ε, στην ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα. Κλείνοντας να πω ότι κανένας εδώ πέρα δεν μπορεί να πιστεύει ότι είναι προσυμφέρον του να αποτύχει η νέα κυβέρνηση για μικροκομματικούς λόγους, διότι η αποτυχία της νέας ελληνικής κυβέρνησης αναπόφευκτα συνεπάγεται την νίκη των δημαγωγών, των αντιευρωπαϊστών δημαγωγών. Σας ευχαριστούμε κύριε Λεύρες. Ο κύριος και το FTD. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να εστιαστώ στην Ελλάδα σήμερα και θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Ντάισελμπλουμ, ο οποίος πριν από δύο μέρες είπε ότι κάνετε λάθος άμα πιστεύετε τη δημοκρατία είναι ε, το ότι ένα εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο τη Ευρωζώνης. Ε, και κύριε Γιούγκερ, εσεί είχατε πει ότι δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατική επιλογή κατά τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και των συνθήκων τη. Αυτά, αυτά χρειάζεται να ξέρουμε, θεωρώ, για την οικονομική αντίληψη τη Ευρώπη και την, για την οικονομία. Καταστρέφουμε τη δημοκρατία εκεί που δημιουργήθηκε, στην Ελλάδα. Έχετε επιτρέψει στην Ελλάδα να μπει σε ένα νόμισμα στο οποίο δεν θα έπρεπε να έχει μπει. Έχετε αφαιρέσει, καθαιρέσει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό όταν έθεσε δημοψήφισμα. Έχετε επιβάλει λιτότητα η οποία έχει πάρει από τον ε, λαό της Ελλάδας τα απαραίτητα για να ζήσει και τώρα ζητάτε οικονομική αλλαγή. Κυριαρχία και δημοκρατία στην Ελλάδα δεν είναι δικά σας για να τα σπαστείτε και να τα πάρετε. Έχουν αρκετά υποφέρει οι ε, Έλληνες. Είναι σαφής ε, η μαχή οι δυνάμεις της Ελλάδας κατά τις ε, δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ζητώ το εξή να σταθούν όρθιοι και στον, στον ελληνικό λαό λέω να είναι τολμηρός γιατί εσείς ιδρύσατε την δημοκρατία και πρέπει τώρα να τη σώσετε πρέπει να επικαλεστείτε το πνεύμα των προπατώρων σας. Να μην ε, λυγίσετε, να μην υποχωρήσετε. Εσείς είσαστε οι πρόσπιστε τη δημοκρατία τώρα. Εσείς είστε το έθνο του Ομήρου, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη. Και αν κρατήσετε τη θέση σας, θα κυριαρχήσετε και θα γίνετε φάρος ελπίδα για όλους μας. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Λεπέν. Παρακολουθούμε την νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα, η οποία προσπαθεί να αμφισβητήσει την καταστροφική πολιτική του Τρόικα. Θα πρέπει να μην μείνει μέσα στο ευρώ και προδώσει αυτά τα οποία είπε εναντίον της λιτότητας, πρέπει να φύγουν από το ευρώ για να εφαρμόσουν τη σωστή πολιτική αλλά η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα προτίμησε το ευρώ και προτίμησε την προδοσία των υποσχέσεών της υπέκυψε στην, στον εκβιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον εκβιασμό της Γερμανίας. Ε, υπό το φως του ελληνικού επεισοδίου οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι είδαν την ασυμβατότητα που υπάρχει ανάμεσα στο ευρώ και τη δημοκρατία από τη μία και το ευρώ και την ευημερία από την άλλη πολύ περισσότερο από ποτέ. Το Εθνικό Μέτωπο θέλει να βγάλει την Γαλλία από την Ευρωδικτατορία, δίνοντας τη Γαλλία το νόμισμά της, τα σύνορά της και αποφεύγοντας την υποχρέωση, την υπερχρέωση, τη λιτότητα και την μαζική ανεργία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Γαλλικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Χαίρομαι που το Συμβούλιο ασχολήθηκε κυρίως με τα θέματα της τρομοκρατίας. Το είχαμε πει μετά το Παρίσι. Και η νέα τραγωδία της Κοπενχάγης υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω δράση. Αν υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι οι απειλές που έχουμε μπροστά μας, κυρίως η απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας. Η κυρία Λεπέν ασχολήθηκε και μετά της Ελλάδας. Σημαντικό θέμα. Εγώ θα ασχοληθώ μετά της Γαλλίας, η οποία είναι ίσως και πιο σημαντική. Χαίρομαι λοιπόν κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέση που πήρατε σχετικά με την Γαλλία. Για τρίτη φορά δυστυχώς η Γαλλία δεν καταφέρνει να τιμήσει τις ανηλυμένες της υποχρεώσεις, τις πιο επίσημα ανηλυμένες. Όπως είπατε είναι υπό ενισχυμένη επίβλεψη πλέον η Γαλλία. Είναι μια θα έλεγα στάση επιφύλαξης και δυστυχώς είναι τεκμηριωμένη. Και από ό,τι κατάλαβα θα έχει μόνο τρεις μήνες για να παρουσιάσει νέες θέσεις, ενώ η ελληνική κυβέρνηση θα έχει έξι μήνες. Ε, θα πρέπει τέσσερα δις να εξοικονομήσει η γαλλική κυβέρνηση, που θα οδηγήσουν σε 16 δις το 2016 και το 2017. Ευχαριστούμε την Ευρώπη γιατί πραγματικά υποχρεώνει μια κυβέρνηση χωρίς θάρρος και χωρίς πλειοψηφία να εφαρμόσει μια πολιτική που θα σώσει τη χώρα. Και τώρα για τον Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε, ο κ. θα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η τελευταία άτυπη συνάντηση των αρχαίων κρατών και κυβερνήσεων έλαβε χώρα με λίγε ώρε μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων. Η κατάσταση στην ε, ανατολή τη Ουκρανία έχει κάπω βελτιωθεί, αλλά η συμφωνία της, του Μίνσκ δεν έχει εφαρμοστεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει εφαρμοστεί. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι έχει δίκιο ο κ. Περχόφστατ. Θα πρέπει να σταματήσουμε να αντιδρούμε κάθε φορά εκ των υστέρων όταν συμβαίνει ήδη κάτι. Θα πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι εκ των εκ των προτέρων για το τι θα συμβεί εάν συνεχιστεί αυτή η τάση και αν δεν εφαρμοστεί η συμφωνία του Μίνσκ. Και αντιστρόφως, τι θα μπορούσε να συμβεί αν από κοινού ακολουθήσουμε άλλο μονοπάτι από αυτό που ακολουθεί προς το παρόν η κυβέρνηση της Ρωσίας. Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι τέτοια που επιβάλλει σαφή λόγια και σαφή γλώσσα και δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στην ομοφωνία, θα πρέπει να υπολογίζουμε και τι θα συμβεί και χρειάζεται λοιπόν σαφής ε, γλώσσα και σαφής κυρώσεις αν δεν τηρηθούν οι συμφωνίες. Και τότε θα πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται και με αυτούς που δεν θέλουν να στρατιωτική λύση και γι' αυτό οπλισμό. Ένα πράγμα θέλω να σας παρακαλέσω σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, να ελέγξετε αν οι βουλευτές του Ρωσικού Κοινοβούλιο ε, που είναι στον κατάλογο των ε, αυτών στον οποίο θα επιβληθούν κυρώσεις θα πρέπει να παραμείνουν. Γιατί ο διακοινοβουλευτικός διάλογος δεν γίνεται ουσιαστικά πλέον και αυτό είναι κρίμα. Σα ευχαριστώ και τώρα για το ECR, του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. το λόγο έχει κύριο Λούκε. Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα σε μια επιστολή ζήτησε παράταση τη πιστοτική βοήθειας και η ερμηνεία είναι ότι η Ελλάδα ζητάει παράταση. Εγώ ε, έχω μια άλλη ερμηνεία, γιατί διάβασα ε, την επιστολή και δεν είδα ακριβή αριθμητικά στοιχεία. Τι ακριβώς μας προσφέρει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά εξοικονομίες για τις δαπάνες που θέλει να κάνει. Ξέρουμε ε, τις συζητήσεις που έγιναν, αλλά δεν ξέρουμε τι θα είναι, ποια θα είναι τα έσοδα, ξέρουμε ποια θα είναι τα δαπάνες. Βελτίωση της φορολογίας και της φοροσυλλογής. Πόσα εκατομμύρια αυτό και δισεκατομμύρια θα σημαίνει για τα ελληνικά ταμεία. Ποιες ε, θα είναι συγκεκριμένες τα έσοδα σε ευρώ. Δεν θα πρέπει να γίνουν άλλες ε, ε, ιδιωτικοποίησεις. Τι θα γίνει με το, την μεταρρύθμιση του συνταξιδοτικού συστήματος. Κύριε Γιούγκερ, βλέπω ότι η Ελλάδα δεν έχει δώσει αριθμητικά στοιχεία, αλλά έχει δώσει πληρωμέ. έχει λάβει πληρωμές. Νομίζω ότι τελικά πέρασε αυτό που ήθελε η Ελλάδα. Ο κύριος Άλμπρεχτ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Πρόεδρε, αξιότιμη συνάδελφοι. Για το PNR είναι σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αρμόδια Επιτροπή, η Επιτροπή ε, παρέπεμψε το θέμα αυτό επειδή θεωρήσαμε ότι ήταν ε, ανισόρροπο το θέμα αυτό και δεν υπήρχε η απαραίτητη αλλαγή πλέον. Δεν μπορώ να δω λοιπόν πώς το Κοινοβούλιο μπορεί να συμφωνήσει με την σημερινή πρόταση που δεν έχει αλλάξει και δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε το, την επιχειρηματολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποφάνθηκε ότι δεν είναι σύνομη η τήρηση τέτοιων αρχείων. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτείνω να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει μια νέα πρόταση. Δηλαδή δεν πρόκειται να προχωρήσει καθόλου το θέμα αυτό. Και τώρα για το EFTD το λόγο έχει η κυρία Μπεγκίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην πρόσφατη συνάντησή τους μίλησαν για το μέλλον της Ελλάδας, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Κανένας δεν βλέπει το πρόβλημα καλύτερα από ότι οι Έλληνες. Οι Έλληνες πρέπει να αποφασίσουν για το μέλλον της χώρας τους. Και όμως εμείς καθόμαστε και συζητάμε το τι λέει το Βερολίνο, το τι λένε οι Βρυξέλλες και πώς αντιδρά ε, κάποια άλλη πρωτεύουσα. Νομίζω ότι δεν μπορεί η μοίρα ενός λαού να είναι στα χέρια των άλλων. Αυτό είναι λάθος. Και από ό,τι φαίνεται ο Πρωθυπουργό της χώρας αναγκάστηκε να δεχτεί τις θέσεις της Γερμανίας και άλλαξε όλες τις θέσεις που είχε. Και φυσικά αυτή ήταν μια προειδοποίηση για τις άλλες χώρες. Μα ποιος είναι ο Γιούγκερ και ποια είναι η Μέρκελ αυτή η, η, αγιατολά της αυθαιρεσίας που θα επιβάλλουν τις απόψεις ε, στην ε, Ελλάδα για να επιβάλλουν αυτές τις θυσίες και τις ε, περικοπές. Η κρίση στην Ελλάδα δεν είναι μια ελληνική κρίση, είναι μια ευρωπαϊκή κρίση, δεν είναι μια οικονομική κρίση, είναι μια πολιτική ε, κρίση. Είναι μια μικρή χώρα η οποία έχει το ΑΕΠ μιας μεγάλης Ιταλικής ή Γαλλικής επαρχίας. Μπορούμε να τη σώσουμε όποτε θέλουμε. Όμως είναι η κρίση μιας Ευρώπης η οποία είναι μίζερη, είναι μια Ευρώπη η οποία δεν θέλει να έχει την πολιτική ε, ε, θέληση. Ελείπουν οι πραγματικοί πολιτικοί αρχηγοί που θα μας βγάλουν από την κρίση. Ο κ. έχει το λόγο η συμφωνία eurogroup κυβέρνηση συριζα ανέλ στην ελλάδα επεκτείνει το μνημόνιο και με την επιτήρηση της τρόικας με άλλο όνομα. η ευρωπαϊκή ένωση δεν αλλάζει. κάθε διαπραγμάτευση με αυτήν είναι απάτη και καταλήγει πάντα σε βαρβαρότητα. ο λαός που μάτωσε θα συνεχίσει να πληρώνει ένα χρέος που δεν οφείλει με εθνικό στόχο τα κέρδη του κεφαλαίου με ιδιωτικοποιήσεις φόρους τσακισμένους μισθούς συντάξεις κοινωνικές παροχές νέα μέτρα για λιτό βίο ακόμα και τα ψίχουλα στην ακραία φτώχεια και η αύξηση του βασικού μισθού αναβάλλονται αν και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και η τρόικα. η κυβέρνηση παρουσιάζει το λαό σαν χειροκροτητή αυτής της πολιτικής αλλά κανείς δεν ξεμπέρδευσε ακόμα με το λαό. καμιά ανοχή κατάρριξη του μνημονίου με ανάκτηση όλων των απολειών διαγραφή του χρέους και αποδέσμευση από την ευρωπαϊκή ένωση. αυτή είναι η πραγματικά αξιοπρεπή στάση του λαού μας που θα ακουστεί δυνατά την παρασκευή στην αθήνα στη μεγάλη συγκέντρωση του κομμουνιστικού κόμματος ελλάδας. Äh, το λόγο έχει ο κύριος Κοντσάλας Πόντς ε, για το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, το ψήφισμα για την τρομοκρατία που έγινε δεκτό από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και οι δηλώσεις του Συμβουλίου κατά της τρομοκρατίας αποδεικνύουν ότι ακολουθούμε τη σωστή διεύθυνση, κατεύθυνση. Ε, νομίζω ότι και στην Ισπανία συμφωνεί και το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία αλλά δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια, θα πρέπει η ενότητα την οποία έχουμε επιδείξει σε επίπεδο τριών θεσμικών οργάνων να γίνει πραγματικότητα. Νομίζω θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και να προωθήσουμε θέματα όπως το PNR, ο κατάλογος των ονομάτων των ταξιδιωτών στις αεροπορικές εταιρείες ευρωπαϊκού τύπου, σεβόμενοι φυσικά πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα προχωρήσει με τα λόγια, θα προχωρήσει με τις πράξεις και δεν εξαρτάται από άλλους. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και πρέπει να θυμόμαστε πάντα τα θύματα της τρομοκρατίας. Η χώρα μου, η Ισπανία, ε, πραγματικά ζητά και μια πλήρη, μια πραγματική ε, ενότητα ενέργειας. Η Πορτογαλία και η Ισπανία ζητούν να υπάρξει μια πραγματική δικτύωση στον τομέα της ενέργειας ε, με την υπόλοιπη Ευρώπη. Κανένας δεν μπορεί να είναι μια ενεργειακή νήσος, αλλά σε καμία περίπτωση ούτε και η Ελλάδα μπορεί να απομονωθεί σοσιαλιστές η κυρία Φερέιρα τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η προσωρινή συμφωνία που επετέφθη για την Ελλάδα είναι πρόσδεκτη, αλλά δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Είναι η απαρχή μιας νέας φάσης που πρέπει να είναι διαφορετική. Ε, στραγγαλίζεται από πολιτικές προσαρμογής, υπερβολικές πολιτικές προσαρμογής ε, η Ελλάδα και η οικονομία, η απασχόληση, η κοινωνία, η εμπιστοσύνη καταρακώθηκαν ε, όπως ε, ο, ο κύριος Ζαν Κλοντιούνκερ αναγνώρισε. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ε, σίγουρα χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, σίγουρα πρέπει να διορθώσει την πορεία της ε, η Ελλάδα, όμως ε, σταδιακά και με ένα δημοσιονομικό περιθώριο που το επιτρέπει. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες σήμερα. Οι εναλλακτικέ λύσεις σε σχέση με την παράλογη πολιτική της λιτότητας υπάρχουν. Και αυτές οι εναλλακτικέ χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένα νέο πρόγραμμα ε, χρειάζεται επικαιροποίηση του προγράμματος. Ε, ας αφήσουμε λοιπόν τις επιδείξεις ισχύω, ας αφήσουμε τα κηρύγματα. Αυτά είναι επικίνδυνα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την επιβίωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ε, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα προγράμματα βασιζόμενοι στα αποτελέσματα και όχι βάσει κοντόφελμου συμφερόντων. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για το ECR κυρία Στίβενς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες ε, παρατηρήσεις. Ε, συνάδελφοι ευρωβουλευτές, σας καλώ την έκθεση του Τίμωθη και το PNR σας ε, καλώ να την προσεγγίσετε με επικοδομητικό τρόπο. Πέρα από δόγματα, να κοιτάξουμε θέματα που πραγματεύεται και να δώσουμε την απαραίτητη ορμή. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό γρήγορα να καταρτήσει εφαρμοστικές διατάξεις για συγκεκριμένες, συγκεκριμένους δείκτες για πιο στοχευμένους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, κατά τα κράτη-μέλη για πιο πολύ εμπιστοσύνη το ένα στο άλλο και πιο εντατική ανταλλαγή απόψεων και λειτουργική συνεργασία μέσω της πόλου. Τέλος, προσβλέπω στην ε, μεταρρυθμισμένη ε, έκδοση της στρατηγικής για την ιστορική ασφάλεια τον Απρίλιο, γιατί η Ευρώπη μπορεί να σημαίνει και να προσφέρει πιο πολύ προστασία και συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει από το EFTD η κυρία, ο κύριος Λουνγκριν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Τούσκο και στον κύριο Γιούνκερ. Ε, συνέχεια τα ίδια ρωτάω, αλλά δεν, άοκνα θα εξακολουθήσω να επαναλαμβάνω αυτά τα ερωτήματα. Τι κάνετε εσείς ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, ε αντιπροσωπεύετε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους ε, που δεν σας έχουν ψηφίσει. Μπορούμε, μπορείτε όμως να αποφασίσετε τι θα γίνεται στη ζωή τους. Ε, Αποφασίζει να περικόπτεται τους μισθούς και τις συντάξεις. Ε, ταυτόχρονα όμως ε, πολλαπλασιάζονται τα μπόνους για τους τραπεζίτες. Έχουμε άπειρα παραδείγματα για αυτά και βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιοι έχουν φόρου ζωής, συντάξεις μόνο και μόνο επειδή παίρνουν τέτοιες λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, θα σταματήσετε εσείς αυτήν την πρακτική Εκεί θα απαρνηθείτε αυτά τα προνόμια όταν εσείς αποχωρήσετε από τη δική σας θέση γιατί τα πληρώνουν όλα αυτά από το πορτοφόλιο τους οι πολίτες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βιλίμσκι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία συζήτηση για το Συμβούλιο μας δίνει την εντύπωση ότι από σύνοδο σε σύνοδο τα πράγματα χειροτερεύουν και πάνε και βρισκόμαστε σε ένα πολιτικό τιτανικό και γενικώ ε, μάζει νερά το πλοίο αυτό. Και δεν καταφέρνουμε να γεμίσουμε, να κλείσουμε τις τρύπες. Μαζική ανεργία σε επίπεδα νερό, ρεκόρ. Το ευρώ δέχεται πιέσεις και τώρα θέλετε να αποφασίζετε άλλο τι θα γίνει με άλλη μια πληρωμή προς την Πελοπόννησο να κατανοήσουμε ότι και αυτά θα είναι χαμένα χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια σφάλματα στην αρχή της. Η κεντρική ρύθμιση, η εποπτεία, η καταναγκαστική εποπτεία και παρακολούθηση. Όποιος θέλει μέλλον στην Ευρώπη θα πρέπει να κάνει μία επαναχώρηση, να κινηθούμε προς την κατεύθυνση, προς την κοινότητα κυρίαρχων εθνών που θα συνεργάζονται και θα σταματήσουν αυτή την ε, καταναγκαστική κεντρική διαμόρφωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ραγγέλ από πλευρά του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα φυσικά να χαιρετήσω τον πρόεδρο του Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τα αποτελέσματα που είχαμε, την όθηση που δίνουν, τη νέα δυναμική που δίνουν μέσα από αυτό το άτυπο Συμβούλιο για τη τρομοκρατία πρώτα απ' όλα. Ήταν σημαντικότατη η πρόοδος, πιστεύω εγώ, και ταυτόχρονα ε, κατοχυρώνουμε το Σέγγεν, είναι θεμελιώδη σημασία, γιατί διαφυλάται την ελευθερία κυκλοφορία. Σε δεύτερο η Ουκρανία κρίνω ότι ε, παρόλα αυτά που έχουν επιτευχθεί υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες και φυσικά το θέμα της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ε, με εστίαση στην Ελλάδα. Θα ήθελα να πω το εξή. Κρίνουμε ότι είναι καλή και λογική αυτή η συμφωνία διότι κατάλαβε η ελληνική κυβέρνηση ότι καταλητική σημασία για την αλληλεγγύη, για την υπέρβαση των προβλημάτων δικαιωμάτων της ε, είναι να ε, συμμορφωθεί με τους κανόνες ε, της Ευρωζώνης και ακολουθεί έτσι ένα ε, δρόμο ε, που οδηγεί, θα οδηγήσει μετά από λίγους μήνες ε, μαζί με κάποιες εγγυήσει σε μια νέα έκβαση. Αλλά είναι ένας δρόμος της ελπίδας και γι' αυτό θα έλεγα ότι με αυτό το άτυπο συμβούλιο νομίζω ότι δημιουργήθηκε μια νέα ελπίδα. Για τους σοσιαλιστές η κυρία Γιώτοβα τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αφαιρθώ στα μέτρα τα οποία ε, θα πρέπει να ληφθούν κατά της τρομοκρατίας. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Δεν έχουμε όμως και μία ανάλυση σε βάθος ε, για το φαινόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα που θα υιοθετήσουμε τη νέα στρατηγική στον τομέα της ασφάλειας χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη θα μπορούν να συνεργαστούν στα πλαίσια της Europol και της Interpol. Απαιτείται αλληλεγγύη, απαιτείται αμοιβαία αναγνώριση των προσπαθειών στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Και θα πρέπει το σύστημα Schengen όχι να το συρρυκνώσουμε αλλά να το αναπτύξουμε. Ε, έχουμε σύνορα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Βουλγαρία, η Ελλάδα κτλ και θέλουμε βοήθεια για να ελέγξουμε τα σύνορα αυτά. Υπάρχει επίσης και υψηλή μεταναστευτική ε, πίεση. Εμείς ε, θα πρέπει ε, να παίξουμε το ρόλο μας, αλλά να μην υπολογίζεται μόνο σε εμά για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των υπολείπων χωρών. Τη διαπραγμάτευση μεταξύ της νέας ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών, όπως πλέον θα πρέπει να συνηθίσουμε να τους προσφωνούμε κατέδειξε με σαφήνεια ότι η ευρωπαϊκή ένωση υποκύπτει στις επιθυμίες της γερμανίας και των φίλων της. ενώ της δόθηκε η ευκαιρία να δείξει ότι ενδιαφέρεται για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών μελών και κατ' επέκταση των πολιτών της απέδειξε απερίφραστα την αγκύλωση στις διαθέσεις της γερμανίας για εκμετάλλευση της κρίσης των χωρών του νότου προς όφελός της. δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σύμφωνα με έρευνα του london school of economics τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού της γερμανίας την τελευταία πενταετία απέφεραν έσοδα στο βερολίνο της τάξης των 80 δις ευρώ ένα γεγονός το οποίο δεν γνωρίζουν οι λαοί της ευρώπης. ας σταματήσει επιτέλους αυτή η εκμετάλλευση και η χειραγώγηση. η ευρωπαϊκή ένωση δεν είναι ιδιοκτησία συγκεκριμένων χωρών. ας προσπαθήσει πρώτα η γερμανική κυβέρνηση να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις της και μετά να κάνει μαθήματα σε άλλους. η ελλάδα βέβαια δεν πρόκειται να παραιτηθεί από το δικαίωμά τη, να διεκδικεί και το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Karas, το έλεξα. Ε, παρακαλώ κυρίες και κύριοι από τον εξώστη, σας παρακαλώ να μην ε, κάνετε φασαρία και δεν επιτρέπονται τα χειροκροτήματα. Κύριε κύριος ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι για κανένα από εμά δεν είναι ικανοποιητικό το ότι γίνεται στο θέμα με Ουκρανία, Ρωσία, ε, Ελλάδα, ε, τρομοκρατία, εξωτερικά σύνορα. Κανείς δεν μπορεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να αποφανθεί και να δώσει μια ικανοποιητική λύση για το μέλλον. Γι' αυτό θα ήθελα στην βασικό σχεδιασμό να πω το εξή. Κανένα θέμα δεν μπορούμε να το δούμε και να το θεωρήσουμε απομονωμένο. Πάντα μιλάμε για το σύνολο της Ευρώπης. Είναι τα δικά μας προβλήματα, όχι τα προβλήματα άλλων. Και η αιτία για όλα αυτά τα ζητήματα, για τα προβλήματα, είναι η παραβίαση του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου και η παραβίαση των κοινών μας αξιών. Και ως εκ τούτου η απάντησή μας θα πρέπει να εστιαστεί στο πώς μπορούμε στην ε, επικράτειά μας πώς μπορούμε στον πυρήνα των αξιών μας να δώσουμε τις σωστές απαντήσεις σε αυτές τις παραβιάσεις. Δεν θα πρέπει να αλλάξουν οι αξίες μας και η νομοθεσία μας λόγω των παραβιάσεων. Όχι. Θα πρέπει τα δικές μας αξίες να δώσουν εμπιστοσύνη και κύρος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και ως εκ τούτου είναι πραγματικά ε, ανήκουστο το γεγονός ότι στην τηλεόραση στην Ελλάδα βλέπω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργό μετά από μια συμφωνία για μια νομική συμφωνία λέει ότι κερδίσαμε μια μάχη αλλά όχι τον πόλεμο. Δεν μπορεί αυτό να οικοδομήσει εμπιστοσύνη. Όταν ένα κυβερνητικό κόμμα αναφέρει τέτοια ζητήματα. Και γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να προσπιστούμε αυτά με τις δικές μας αξίες, αλλά διακόπτει ο Πρόεδρος, δυστυχώς, το λόγο τώρα έχει για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες η κυρία Κέγγε. Ε, Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να υποστηρίξουμε με συντονισμένο τρόπο την προσπάθεια όλων των χωρών να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία. Πρέπει να ευνοήσουμε τις διαδικασίες ειρήνευσης για να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας και την κοινωνία μας και την ασφάλειά μας αλλά και τους άλλους λαούς. Απαιτείται μια σφαιρική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας δεν θα πρέπει να περιοριστούμε ε, στην αντιμετώπιση των πιο κοντινών σειράξεων όπως τη Λιβύη. Θα πρέπει όμως να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτό το παγκόσμιο δίκτυο της ε, τρομοκρατίας. Ξεχνάτε τι συμβαίνει στην Βόρεια Νιγηρία με τον Μπόκο Χαράμ. Την ξεχνάμε την κρίση αυτή, την κρύβουμε. Τα ίδια προβλήματα έχουμε με τους Ντάες στην Λιβύη και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Στις βαρβαρότητες αυτών των ομάδων δεν πρέπει να μείνουμε αδιάφοροι. Σας ευχαριστώ από το ΕΛΚ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Σούιτσα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που εκπροσωπούνται τα τρία θεσμικά όργανα από τους τρεις προέδρους και χαίρομαι διότι έχουμε πλέον ομοφωνία σε σχέση με την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών. Αυτό που ακούσαμε στο τελευταίο Συμβούλιο ε, σχετίζονται με την αξιοπρέπεια, με τη ζωή την ίδια των πολιτών. Αυτό θα πρέπει να διαφυλάξουμε. Αυτό ήταν ε, το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα ε, ε, ήταν ε, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση και στη συνέχεια το επενδυτικό σχέδιο. Δηλαδή πρώτα συζητήθηκαν τα προβλήματα και στη συνέχεια οι λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Θα πρότεινα λοιπόν να προωθήσουμε την Ενεργειακή Ένωση, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την Ενεργειακή Ένωση για να μπορέσουμε να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ε, αντιμετωπίζει η Ελλάδα, ε, τα προβλήματα που έχουμε με τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, τα προβλήματα με την Ουκρανία. Πολύ καλό που συμφώνησαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, όμως στην πράξη θα δυσκολευτούμε να λύσουμε το πρόβλημα της Ουκρανίας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στο Κοινοβούλιο για να μας ενημερώσετε. και Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό που πολλοί εδώ υποστηρίζουμε, δηλώνουμε αλληλέγγυη σε με την ε, ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό που αντιμετώπισε τόσες ε, δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Ε, πολύ συντηρητικοί μετά τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια ε, μιλούσαν σαν να έπρεπε να πληρώσει ο ελληνικός λαός ε, για το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών. Το αντίθετο, έχουμε χρέος να βοηθήσουμε την Ελλάδα για να αναδιατάξει το μη βιώσιμο χρέος της ε, για να διορθώσει το φορολογικό της σύστημα για να τονώσει και πάλι την οικονομική δραστηριότητα. Εγώ Λυπάμαι διότι με τις δηλώσεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, νομίζουμε ότι τελειώνει η δημοκρατία στα όρια της συνθήκης λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να έχουμε αυτές τις έμονες ιδέες, ε, να είμαστε δέσμοι αυτών, ε, να ξεκινήσουμε σε αυτήν τη νέα φάση. Διακόπτει ο Πρόεδρος, ο κύριος Σβέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το τελευταίο άτυπο συμβουλίο ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Ένα από τα αποτελέσματα, ένα από τα συμπεράσματα είναι ότι το Eurogroup ενέκρινε το νέο σχέδιο μεταρρυθμίσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Ελπίζω ο κ. Τσίπρας να συνεχίσει να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις. Ελπίζω να ενισχύσει τον προϋπολογισμό και ελπίζω η Ελλάδα να ξεπληρώσει τα όσα της δώσαμε. Η Ελλάδα έλαβε πολλά για τις μεταρρυθμίσεις της τα τελευταία χρόνια. Και πληρώνει μικρότερα από εσά σε σχέση με το ΑΕΠ της, ε, σε σχέση με τη Σλοβενία ή με άλλες χώρες. Εγώ θεωρώ ότι φτάνουν, ε, φτάνει η υποχωρητικότητα. Δεν ε, δούλεψε η απειλή της ελληνικής εξόδου. Κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να υπάρξει καμία καταστροφή. Το Eurogroup είναι πολύ ισχυρό σήμερα λοιπόν και θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. να Έχουμε τέσσερα παραπάνω μέλη και δεν έχουμε χάσει κανένα μέθαμα. μέλη. Η κυρία Φραζίκοβα. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολύ δύσκολα προβλήματα και σε εσωτερικό επίπεδο και σε εξωτερικό. Οι τραγωδίες στη Δανία και στη Γαλλία και οι κίνδυνοι που δημιουργήθηκαν και εδώ στο Βέλγιο πρέπει να μας οδηγήσουν στο να ε, πάρουμε επιτέλους κάποια μέτρα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πιεστεί το Κοινοβούλιο για να δεχθεί ε, την νομοθεσία για το PNR. Αντίθετα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντα ε, των πολιτών. Τώρα, για την Ελλάδα. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, κανένας δεν θα ήθελε να είναι στη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι πολύ απαιτητική η κατάσταση και πάρα πολύ δύσκολη. Και θα πρέπει να ζητήσω και, ε, και από τους Έλληνες πολιτικούς να δείξουν αλληλεγγύη ε, και στους υπόλοιπους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Σλοβακία, σαν παράδειγμα, έχουμε ανάγκη και θέλουμε βοήθεια και από την ελληνική κυβέρνηση αν αυτό χρειαστεί. Ο κύριος Γιούνκερ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, όπως και στο Συμβούλιο στις 12 Φεβρουαρίου. Θα απαντήσω σε κάποιες παρατηρήσεις γύρω από τα θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να συγχαρώ τον κύριο Μορέλ, Γάλλος σοσιαλιστής, γιατί είπε ακριβώς τα αντίθετα αυτά τα οποία λέγει η κυβέρνησή του, σοσιαλιστική, καθημερινά. Να τον ε, συγχαρώ επίσης και για την αίσθηση χιούμορ που έχει. Είπε ότι είμαστε πολλοί που συζητάμε. Πού είναι οι πολλοί που τους είδατε. Ε, πραγματικά έχετε αναπτυγμένη αίσθηση χιούμορ κύριε Μορέλ. Τρίτον, θα του πω, όπως και σε πολλούς άλλους, ότι εγώ ποτέ δεν είπα ότι οι εκλογές είναι ένα ουδέτερο συμβάν. Είπα εγώ κάτι το οποίο έχει μια απλή λογική, ότι τα εκλογικά αποτελέσματα δεν αλλάζουν τις συνθήκες. Αυτό είπα. Η Ελλάδα πήρε μια απόφαση σαν κυρίαρχη χώρα και σέβομαι εγώ τα αποτελέσματα της λαϊκής έκφρασης. Περισσότερο από άλλους το σέβομαι αλλά ταυτόχρονα η Ελλάδα και η ελληνική ψήφος δεν έχει σαν αποτέλεσμα μέσω απλά των αποτελεσμάτων των εκλογών να αλλάξουν οι συνθήκες και ε, οι συμφωνίες που έχουν γίνει. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εκλογές στην Εστονία. Τον Απρίλιο θα έχουμε εκλογές στη Φιλανδία. Ε, τι θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή πιστεύετε ότι μετά από κάθε εκλογική διαδικασία θα πρέπει να αμφισβητούμε τις συνθήκες και τους κανόνες. Θα σκοτώσουμε την Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο. Παρακαλώ μην τα λέτε αυτά γιατί πρέπει να φανούμε ορθολογικοί και ε, να σεβαστούμε την κοινή λογική. Γιατί πολλές φορές αυτό δεν φαίνεται να το κάνουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Ασκήθηκε πάρα πολύ κριτική εις βάρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον τελευταίο καιρό θα πρέπει να πω. Πολλές φορές ζητούσαμε από τους δημοσιογράφους ότι τους να γράψουν αυτά τα οποία πίστευαν οι κυβερνήσεις τους. Είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εμπλακεί με απαράδεκτο τρόπο στη συζήτηση για την Ελλάδα. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, της είχε ασκηθεί στο παρελθόν κριτική ε, ότι δεν είχε εμπλακεί ε, σωστά και σε βάθος στα θέματα αυτά. Και τώρα ασκούμε κριτική πάλι στην ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ανακατεύεται σε εισαγωγικά με ό,τι έχει σχέση με την νομισματική και την οικονομική πολιτική. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει σαν αποστολή να διαιρεί την Ευρώπη. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει μια ενωτική αποστολή εκεί όπου αμφισβητείται η Ένωση. Και ε, η ενότητα της Ευρώπης, ε, η καταδίκη της, των πιθανών ρήξεων είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάναμε αυτό το οποίο απλά έπρεπε να κάνουμε. Και αν δεν το είχαμε κάνει, δεν θα είχε υπάρξει πάρα πολύ απλά συμφωνία ε, πάνω στην Ελλάδα. Τώρα, για τα υπόλοιπα. Γιατί μιλάμε πάντα για το ότι κάποιος πέρασε το δικό του. Αν περνάει κάτι κάποιος, σημαίνει ότι καταπιέζει τους άλλους. Το θέμα είναι σήμερα αν πέρασε το δικό της η Ελλάδα ή, το Eurogroup. Τι, τι νόημα έχουν αυτές οι συγκρίσεις, αυτές οι συζητήσεις. Δεν έχει κανένα νόημα στην Ευρώπη περνάει η ευρωπαϊκή λύση. Περνάει αυτός που βρίσκει ευρωπαϊκές λύσεις. Κανείς δεν καταπιέζει τον άλλον. Είναι πολιτικές ανοησίες αυτές. Μέσα μετά από κάθε απόφαση να ελέγξουμε δηλαδή ποιος πέρασε το δικό του. Κανείς στην Ευρώπη δεν χρειάζεται να πέρασε το δικό του. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή σκέψη. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο Πρόεδρος Τούσκ. Thank Ευχαριστώ. Δύο σύντομες παρατηρήσεις μόνο, Πρόεδρε. Πρώτον, για την Ουκρανία. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε ο Γκίφι Φεχόφστατ. Θα πρέπει να είναι πιο προδραστική η πολιτική μας, η στρατηγική μας. και συμφωνώ δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε ε, την ε, στρατηγική με κοινέ δηλώσεις. Ξέρετε φυσικά τι εννοώ όταν μιλάω για νέα στρατηγική. Ομο... Ομονοούμε και αυτό είναι καλό γιατί αυτό είναι η πρώτη και βασικότερη προϋπόθεση για να κάνουμε οτιδήποτε. Χρειαζόμαστε τη στρατηγική, αλλά χωρίς τη συνένεση δεν θα τελεσφορήσουν οι προσπάθειές μας. Ο πρώτος λόγος είναι ένας πολύ πρακτικός λόγος. Όλοι οι δράσεις που αναλαμβάνουμε, οι κυρώσεις, παραδείγματος χάρη, προϋποθέτουν συνένεση στο Συμβούλιο. Δεν είναι ότι για ιδεολογικούς λόγους οραματίζουμε, πρέπει όλοι να ομονοούμε. Όχι, για πρακτικούς λόγους δεν μπορούμε διαφορετικά. Τη χρειαζόμαστε τη συνένεση. Δεύτερον, γιατί μιλάμε διαρκώς για την ενότητα, για την συνένεση. Πιστεύω πραγματικά και ελπίζω να μην σας εκπλήσει αυτό πως ένας από τους βασικότερους στόχους που έχει ο πρόεδρος Πούτιν είναι το διέρη και βασίλευε. Αυτό σε σχέση με ε, όλες τις δυτικές χώρες. Γι' αυτό μου έχει γίνει έμονη ιδέα να συμφωνούν μεταξύ τους τα κράτη-μέλη και με την ε, ευρύτερη ε, προοπτική βεβαίως. Το Μάρτι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να συζητήσουμε διεξοδικότερα στην πράξη ποια στρατηγική θα δρομολογήσουμε, όμως δεν έχει κανένα νόημα αυτό εάν δεν ε, υπάρχει ομοθυμία. Δεύτερον, για την Ελλάδα. Δεν συζητούμε εδώ για ιδεολογίες για ένα πόλεμο που κάνουν κάποιοι κατά της Ελλάδας. Εγώ δεν πιστεύω ότι θέλει να είναι μόνιμος ε, ταραχοποιός ε, στην Ευρώπη η Ελλάδα. Το θέμα μας είναι βοήθεια. Η βοήθεια που χρειάζεται η Ελλάδα, τα λεφτά που χρειάζεται η Ελλάδα δεν είναι τίποτα αφηρημένο. Αφήστε που δεν έχουμε και χρόνο. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται ανάμεσα σε κράτη-μέλη, σε εταίρους, σε φίλους. Η πρώτη δημόσια δήλωση που άκουσα από τον Πρωθυπουργό Τσίπρα μετά τις εκλογές ήταν πως η Ελλάδα θέλει να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Και ότι χρειάζεται η Ελλάδα τη βοήθειά μας. Από πλευράς της Ρωσίας ή της Κίνας δεν άκουσα καμία συγκεκριμένη πρόταση για να βοηθηθεί η Ελλάδα. Η μόνη δυνατότητα είναι να τη βοηθήσουν τα μέλη της Ευρωζώνης, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ενδεχομένως. πρέπει να συσπηρωθούμε και να δράσουμε μαζί και να μην αφήσουμε κανέναν να μας διχάσει. Νομίζω πως αυτό πλέον είναι ξεκάθαρο στο μυαλό των πολιτών στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε καλή συνεργασία και όχι τσακωμούς στην Ευρώπη. Όχι να τρογόμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια προβλήματα ε, θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό ένα στον άλλον στις συζητήσεις που γίνονται. Όταν ναι, νιώθει κανείς προσβεβλημένος τότε δυσχεραίνεται αυτόματα και η διαδικασία εξέβρεσης λύσης. Α συζητήσουμε ανοιχτά και α μην προσβάλλουμε οι μεν του δε. Αυτή την πρόταση κάνω εγώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε του Συμβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρίες και κύριοι για το γεγονός ότι δεχτήκατε να τηρήσουμε αυστηρά τα χρονικά όρια. Σήμερα δεν θα μπορούσε να υπάρξει διαδικασία catch the eye γιατί είμαστε υπό εξαιρετική πίεση σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να δείξετε κατανόηση για το γεγονός ότι ούτε μπλε κάρτες αλλά ούτε και catch επετράπηκε. Και έτσι ολοκληρώθηκε η σχετική συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ.